από τους μη εγγεγραμμένους έλαβα αίτημα για ορισμό σε επιτροπή θα δημοσιευτεί στα πρακτικά. Εάν μέχρι την έγκριση των πρακτικών δεν έχει υπάρξει κάποια αντίρρηση, τότε επιβεβαιώνεται αυτός ο διορισμός. Τετάρτη.